Βρετανών, παραδείγματο χάρη, που έχουν ε, εξοχικέ κατοικίε στην Ισπανία ή σε άλλα μέρη και το δίκαιο το οποίο διέπει τέτοιε περιπτώσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και ολοκληρώνουμε τώρα την κοινή συζήτηση για τα θέματα αυτά. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο το μεσημέρι στι 12. Και με βάση την αίσια διάταξη περνάμε στο επόμενο σημείο που είναι η έκθεση της κυρίας Αντονέσκου που αφορά το δικαίωμα πρόσβαση σε δικηγόρο κατά την ποινική διαδικασία και το δικαίωμα επικοινωνία μετά τη σύλληψη. Κυρία Αντωνέσκου, τέσσερα λεπτά. Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχουμε φτάσει στο τέλος μιας μακράς διαδικασίας η οποία ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πρότασή τους για το δικαίωμα πρόσβαση σε δικηγόρο. Χαίρομαι διότι η Επίτροπος κυρία Ρέντιν είναι εδώ. Χαίρομαι και την ευχαριστώ διότι έχει συνεργαστεί στενά μαζί μας και μας έχει στηρίξει καθ' όλη τη διάρκεια της ε, διαδικασίας διαπραγμάτευσης η οποία ήταν εξαιρετικά περίπλοκη και δύσκολη. Θέλω να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους από τις άλλες πολιτικές ομάδες για τη συνεργασία τους και για τη συνέπειά τους. Το αποτέλεσμα είναι προϊόν ομαδικής δουλειάς δεν θα μπορούσαμε να είχαμε υιοθετήσει τόσο στέρεα θέση στις διαπραγματεύσεις διαφορετικά. Και γι' αυτό σήμερα έχουμε ένα εξαιρετικά ποιοτικό κείμενο. Θέλω να ευχαριστήσω τις διάφορες προεδρίες του Συμβουλίου που συμμετείχαν στο εγχείρημα αυτό και κυρίως την Ιρλανδική Προεδρία η οποία μας επέτρεψε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Με την υιοθέτηση των δύο πρώτων μέτρων του οδικού χάρτη για το δικαίωμα πρόσβαση σε δικηγόρο στην ποινική διαδικασία και για το δικαίωμα επικοινωνίας μετά τη σύλληψη. Μετά από αυτά ε, ε, υιοθετούμε το πιο σημαντικό ε, στοιχείο αυτού του οδικού χάρτη, την πρόσβαση σε επαρκή υπεράσπιση. Τα νομικά δικαιακά συστήματα διαφέρουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν διαφορετικές επιπτώσεις και στην πράξη ε, πρακτικές επιπτώσεις. Όλα αυτά όμως δεν θα πρέπει να, εμποδίζουν την αμοιβαία αναγνώριση. Παρόλο που υπάρχουν κοινέ αρχές ε, που προσδιορίζονται από τον ε, χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων και από άλλα κείμενα και παρόλο που προβλέπεται η βοήθεια από δικηγόρο παντού, η κατάσταση διαφέρει από χώρα σε χώρα. Θα πρέπει να εγγυηθούμε τα βασικά αναγνωρισμένα δικαιώματα και να έχουμε επαγγελματική ε, νομική αρρωγή έτσι ώστε να μπορεί κάθε κατηγορούμενος να ασκεί τα δικαιώματά του. Ε, μιλούμε για διαδικαστικά ε, δικαιώματα και θα πρέπει να γίνουν αυτά πραγματικότητα. Είναι βασικό αυτό για να υπάρχει δικαιοσύνη στο σύστημα. Το να προβλέπετε δικηγόρες στη ποινική διαδικασία και να προβλέπετε επικοινωνία κατά τη στιγμή της σύλληψης είναι ε, στοιχεία εξαιρετικά σημαντικά. Η Ευρώπη είναι ένας χώρος ασφάλειας ε, και δικαιοσύνης. Οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να είναι σίγουροι ότι τα δικαιώματά τους γίνονται απολύτως σεβαστά και δεν καταστρατηγούνται σε καμία περίπτωση όταν ταξιδεύουν θα εάν δεν τους προσφέρεται εύκολη πρόσβαση σε δικηγόρο, τότε η υπεράσπιση στην ποινική διαδικασία θα παραμείνει στη σφαίρα του θεωρητικού. Ε, θα έχουμε νομική συνδρομή από τη στιγμή κατά την οποία οι αρμόδιες αρχές ανακοινώνουν στους, ε, στα άτομα αυτά ότι είναι ύποπτα για τη διάπραξη ενός ποινικού κολάσιμου αδικήματος. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε αυτή την έκθεση η οποία θα εγγυάται τις, τους βασικούς κανόνες που θα εφαρμόζονται στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οδηγία αυτή αποτελεί πολύ σημαντική πρόοδο. Θα διευκολύνει τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα δώσω το λόγο και πάλι στην κυρία Ρέντινγκ που αντιπροσωπεύει την Κομισιόν. Σας ευχαριστώ. Μιλάμε για το κείμενο της πρόσβασης, για το δικαίωμα μάλλον, ε, της ε, πρόσβασης δικηγόρο στη ποινική διαδικασία και το δικαίωμα επικοινωνίας μετά τη σύλληψη. Θα είναι μια μεγάλη στιγμή όταν εγκριθεί αυτό το κείμενο, γιατί θα δείξει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υπερασπίζει τα ατομικά δικαιώματα. Και θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια την κυρία Αντωνέσκου, γιατί όχι μόνο ήταν δύσκολη η δουλειά που έκανε, αλλά έπρεπε να δείξει και ε, μεγάλη διπλωματία για να υπάρξει συμφωνία και μαζί με τους σκιώδεις εισηγητές κατάφερε να σταθεί στο ύψος των φιλοδοξιών αυτής της σημαντικής οδηγίας είναι εν τέλει μια ένα επίτευγμα για το οποίο το Κοινοβούλιο μπορεί να είναι περήφανο. Θα ήθελα επίση, κυρία Εισηγήτρια, το έκανε ήδη, να συμπεριλάβουμε στα συγχαρητήριά μας και την Ιρλανδική Προεδρία, διότι με βάση την εργασία των προηγούμενων Προεδριών διαπραγματεύτηκαν πολύ σκληρά ώστε να ολοκληρωθεί η εργασία αυτή και να επιτευχθεί καλή συμφωνία. Λίγο παραπάνω από δύο χρόνια έχουν περάσει μετά από την υποβολή αυτής μας της πρότασης τον Ιούνιο του 2011 και χάρη στην αφοσίωση και το πνεύμα ε, συμβιβασμού από όλες τις πλευρές επετεύχθη συμφωνία. Γνωρίζω πως οι συζητήσεις δεν ήταν πάντοτε εύκολες, ήταν δύσκολο να βρεθούν συμβιβαστικές, για παράδειγμα για τις εξαιρέσεις ή για τις ε, αλλά έχουμε ένα κείμενο τώρα το οποίο είναι στο ύψο των περιστάσεων και είναι και συμβατό με τις αποφάσεις του, Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Για μένα η πρόσβαση σε δικηγόρο είναι ο πυρήνας των διαδικαστικών δικαιωμάτων, αλλά και ο πυρήνα. των όσων περιμένουν οι πολίτες αλλά και οι νομικοί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 8 ε, εκατομμύρια υποθέσεις γίνονται κάθε χρόνο, κρίνονται κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το δικαίωμα στην υπεράσπιση είναι ένα βασικό στοιχείο για μια δίκαιη δίκη. Ε, με αυτή την οδηγία οι πολίτες θα έχουν ε, την ε, δικαίωμα να ανακρίνονται με παρουσία δικηγόρου. Όταν κάποιος ύποπτος συλλαμβάνεται θα έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με την οικογένειά του. Αν βρίσκεται εκτός της χώρας του θα έχει το δικαίωμα να έχει επαφή με το προξενείο της χώρας του. Και πάρα πολύ σημαντικό είναι επίσης ο εμπιστευτικός χαρακτήρας των, των επαφών και η επικοινωνία επιθυμία ενός υπόπτου με έναν δικηγόρο θα πρέπει να γίνεται σεβασλίζεται η άσκηση του δικαιώματος της υπεράσπισης. Ε, οι εξαιρέσεις είναι πολύ περιορισμένες ε, και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις γίνονται, ε, μάλλον χορηγούνται, όπως πούμε στην περίπτωση γεωγραφικής απομάκρυσης ή απόστασης θα υπάρχει δυνατότητα νομικής συμβουλής, συνδρομής εκεί όπου έχει γίνει η σύλληψη αλλά και εκεί όπου εκδόθηκε το ένταλμα σύλληψης. Η διπλή αυτή εκπροσώπηση είναι μια μεγάλη καινοτομία που εισάγεται από αυτή εδώ την οδηγία και θα εξυπηρετήσει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Θα αγγιηθεί την εφαρμογή ε, αυτών των δικαιωμάτων στην πράξη. Τώρα βεβαίως θα πρέπει να εξετάσουμε και την εφαρμογή αυτής της οδηγίας που θα είναι πολύ ουσιαστική για τον σεβασμό και τη συνοχή καθώς και με την πρακτική εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας όπως για παράδειγμα του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Η οδηγία λοιπόν αποτελεί μια σημαντική καθοριστική συμβολή στην ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης που χρειάζεται ώστε να εφαρμοστεί το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα ε, Εντέλμα σύλληψης ή αμοιβαία αναγνώριση των ευρωπαϊκών εντολών εν γέννη. Θα πρέπει λοιπόν να μετά την ολοκλήρωση και την έγκριση αυτής της ε, έκθεσης ε, θα φροντίσουμε ώστε η ολόκληρη οδηγία να μεταγραφεί στα δίκαιο όλων των κρατών μελών και θα εξετάσουμε στενά πώς θα λειτουργήσουν τα πράγματα στην πράξη και σε έφθετο χρόνο θα υποβάλουμε έκθεση που θα αξιολογεί την εφαρμογή επιτόπου. Είμαι πολύ υπερήφανη για το τι κάνουμε εδώ και για το τι έχουμε πετύχει στον τομέα των διαδικαστικών δικαιωμάτων. Θυμηθείτε, έχουμε την οδηγία για την ε, διερμηνία και τη μετάφραση, οδηγία για το δικαίωμα στην ενημέρωση ε, και στην πληροφόρηση και τώρα οδηγία για πρόσβαση σε δικηγόρο, ενώ παράλληλα έχουμε ε, δουλέψει για την οδηγία περιθυμάτων που υιοθετήθηκε πέρσι και που εξασφαλίζει πως τα θύματα θα έχουν ε, ε, μεταχείριση, θα τη χάνουν μεταχείριση με σεβασμό, θα ενημερώνονται, θα προστατεύονται και θα έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη, ενώ θα μπορούν δραστήρια να συμμετέχουν στις ποινικέ διαδικασίες. Βήμα το βήμα λοιπόν ενισχύουμε τον Ευρωπαϊκό Χώρο Δικαιοσύνης και το κράτος δικαίου το οποίο δένει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να ολοκληρώσουμε το έργο μας στο πεδίο των διαδικαστικών δικαιωμάτων σκοπεύει η Κομισιόν να υποβάλει μέτρα όσον αφορά το τεκμήριο αθωότητας, ιδιαίτερη ασφάλεια για υπόπτους ή κατηγορούμενους που είναι παιδιά, ε, καθώς και για την νομική συνδρομή. Σκοπεύω αυτό να σας το παρουσιάσω ήδη μέσα σε αυτό το φθινόπωρο. Σας τονίζω ακόμα μια φορά το μεγάλο σεβασμό που τρέφω για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνομοθέτη στον τομέα της, ε, του ποινικού δικαίου. Είναι ένα μεγάλο βήμα που κάνουμε τώρα και θα είναι πολύ σημαντικό επίσης νομίζω να πούμε στους πολίτες μας κατά τη διάρκεια των της προεκλογικής για το Ευρωκοινοβούλιο να ενημερώσουμε γι' αυτό το κομμάτι της δράσης μας και τις επιτυχίες που έχουμε εδώ και που έχει ε, διεκπαιρεώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο συνομοθέτης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Επίτροπε και για την αναγνώριση από πλευράς της Κομισιόν. Θα δώσω τώρα το λόγο στους ομιλητές που παρεμβαίνουν στο όνομα της ομάδας τους. Καταρχήν η κυρία Ματιού. για 1,5 λεπτό. Ο πρόεδρος διακόπτη, συγγνώμη, σας διακόπτω γιατί Καταρχήν πρέπει να ακούσουμε την νομοδότηση της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων, τον κύριο Άλμπρεχτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο. Ως ε, εισηγητής ε, της Νομικής Επιτροπής ε, θέλω να σας ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω την Επίτροπο κυρία Ρέντινγκ και την εισηγήτρια την κυρία Αντωνέσκου για την εξαιρετική δουλειά που έκανε και για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε. Πιστεύω ότι ειλικρινά καταλήξαμε σε ένα καλό αποτέλεσμα και αυτό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τους πολίτες της Ευρώπης, ούτως ώστε να έχουν ε, ομοιόμορφη προστασία ε, σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό να είναι δεσμευτικό. Είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα. Πιστεύω ότι πρέπει να ακολουθήσουν και άλλα βήματα και τα επόμενα βήματα είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να κάνουμε στη συνέχεια, όπως είναι ε, η δικαστική αρρωγή, η εμβαία αναγνώριση ε, μέτρων, ε, ε, η διενέργεια δικονομικών πράξεων. Πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να υλοποιήσουν στη συνέχεια αυτά τα δικαιώματα, ούτως ώστε να μπορέσουμε μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσουν σε ακόμη καλύτερη κατάσταση για τους πολίτες. Ευχαριστώ. Τώρα δίνω το λόγο στην κυρία Ματιό, εξ ονόματος του ΕΛΚ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Αντωνέσκου για την επιμονή της και για ε, το ότι επιθυμούσε σφόδρα τη συνένεση. Τη χρειάστηκαν δύο χρόνια, αλλά τα κατάφερε να φτάσουμε σε συνένευση και να έχουμε ένα πολύ ισορροπημένο κείμενο. Πρόκειται για μια μεγάλη νομική μεταρρύθμιση μετά το δικαίωμα ε, στη μετάφραση. Σήμερα και το δικαίωμα στην ενημέρωση. Σήμερα έχουμε το δικαίωμα στην πρόσβαση σε δικηγόρο για όλους τους πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ μεγάλο βήμα προς μια Ευρώπη ε, που θα είναι χώρος δικαιοσύνης για όλους τους πολίτες. Είναι ισορροπημένο το κείμενο. Όλοι λοιπόν θα, θα μπορούν να έχουν ε, σύμβουλο νομικό ο οποίος ε, θα τους συμβουλεύσει για την υπεράσπιση τους Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ο ρόλος του δικηγόρου διευρύνεται έτσι ώστε να είναι αυτός όπου θα εγγυάται την δίκαιη δίκη. Βεβαίως μπορεί να υπάρξουν απαρεκκλήσεις προσωρινές με πολύ περιορισμένο χρονικό περιθώριο σε περιπτώσεις καταπολέμησης τρομοκρατίας. Οποιοςδήποτε είναι ύποπτος ε, και καταδιώκεται θα μπορεί ε, από τη μία ε, η δικαιοσύνη να επιλαμβάνεται και από την άλλη τα δικαιώματά του να προστατεύονται. Θα έπρεπε να ήταν η πρόταση πολύ πιο ε, νομική, να μην μείνουμε στο θεωρητικό στάδιο, αλλά να υπάρξει πρόβλεψη και για πόρους μέσα στο κείμενο, για να μην παραμείνουμε μόνο στη θεωρία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος των Σοσιαλιστών, η κυρία Γκυγιόν, παρακαλώ. Κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, αύριο θα ψηφίσουμε αυτή την οδηγία για το δικαίωμα πρόσβαση σε δικηγόρο. Φτάνουμε λοιπόν σε ένα ενισχυμένο κοινό κατόφλι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάτι το εξαιρετικά σημαντικό. Και βεβαίω ε, αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Θα ενισχυθεί η νομική ασφάλεια των διαφόρων συστημάτων. Ε, αυτό το κείμενο το δουλεύουμε εδώ και δύο χρόνια τουλάχιστον και θα έχουμε και πράγματι θα κάνει πραγματικότητα το δικαίωμα στη δίκαιη δίκη. Διασφαλίζεται, εξασφαλίζεται το δικαίωμα της απόρριτης επικοινωνίας με το δικηγόρο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να κατοχυρωθεί το δικαίωμα της υπεράσπισης Βεβαίως όλοι θέλουμε τις ελάχιστες δυνατές παρεκκλήσεις και εξαιρέσεις και από τη στιγμή που πρόκειται για συμβιβασμό ε, λάβαμε υπόψη ορισμένες εθνικές ιδιαιτερότητες. Ωστόσο ε, πλαισιώνεται αυστηρά κάθε είδους παρέκκληση. Το δικαίωμα πρόσβασης στο δεσιτική χώρο ε, θα πρέπει να συμπληρώνεται από το δικαίωμα στη δωρεάν νομική συνδρομή ή αρρωγή για να είναι ολοκληρωμένο. Και γι' αυτό σας καλώ κυρία Επίτροπε να παρουσιάσετε το ταχύτερο δυνατό πρόταση προς αυτή την κατεύθυνση έτσι ώστε η δικαιοσύνη να γίνει λιγότερο άνηση στην Ευρώπη ε, σήμερα. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ εξ του Άλντε, η κυρία Λάτφορντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήμουν εισηγήτρια για το, την πρώτη έκθεση για τα δικονομικά δικαιώματα, το δικαίωμα στη μετάφραση και στη διερμηνία. Επομένως γνωρίζω πολύ καλά τα θέματα αυτά. Αυτό το κείμενο είναι πιο σημαντικό από τα δύο προηγούμενα. Θα πρέπει να κάνουμε όλα τα βήματα του οδικού χάρτη έτσι ώστε να ανέβει ο πύχης ε, στην ευρωπαϊκή επικράτεια και να φτάσουμε επιτέλους στην αμοιβαία αναγνώριση. Έχουν περάσει 10 χρόνια από το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης και θα πρέπει ε, να προστατεύσουμε όλα αυτά τα δικαιώματα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Αντωνέσκου, να την χαρώ θερμά επίσης θα πρέπει όλα αυτά να ισχύουν για τους υπόπτους, για όλους τους κατηγορούμενους, είτε ε, τους... Ε, ε, έχει επιβληθεί ποινή στερητική της ελευθερίας είτε όχι το κράτος μέλος θα πρέπει να ε, κάνει βήματα έτσι ώστε οι εναγόμενοι να είναι σε θέση να ασκήσουν το δικαίωμα ε, τους να έρθουν σε επαφή με δικηγόρο. Και όπως και το ανέφερε η Αντιπρόεδρος κυρία ε, Ρέντιν, η διτή εκπροσώπηση ε, και στις δύο πλευρές της διαδικασίας είναι πολύ σημαντική στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Εγώ θα ήθελα το Ηνωμένο Βασίλειο να υιοθετήσει αυτή την οδηγία με την κυρία Ντονέσκου. Ε, την ευχαριστώ άλλωστε και τους υπόλοιπους ε, σκιώδες εισηγητές διότι επέδεξαν ευελιξία έτσι ώστε να υπάρχουν και προβλέψεις για το common law, το κοινό δικαιακό σύστημα του Ηνωμένου Βασίλειου ελπίζω πραγματικά η κυβέρνηση της χώρας μου να επιλέξει το opt-in και να ενσωματώσει αυτή την οδηγία η οποία μας ταιριάζει. Και θέλω να τονίσω και την ανάγκη να αντιμετωπιστεί επιτέλους αυτό το σκάνδαλο της τόσο μεγάλης ε, κράτησης πριν από τη διεξαγωγή της δίκης. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος των συντηρητικών ο κύριος e, Ευχαριστώ. Πρόεδρε, μιλάμε για μια πολύ, ένα πολύ σημαντικό νομοθέτημα για το οποίο θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια αλλά να ευχαριστήσω και την Νομική Επιτροπή για τις πολύ ενδιαφέρουσες τροπολογίες και αυτές τις τροπολογίες θέλω να σχολιάσω εντάχει. Υπάρχει μια τροπολογία, η 11, η οποία περιορίζει στο πεδίο ελέγχου για μια σύλληψη αν υπάρχει ε, ενδείξεις ότι κάποιος ε, ύποπτος ε, παρενοχλείται. Αλλά πώς μπορεί κανείς να αποδείξει ότι παρενοχλείται κάποιος ενώ συλλαμβάνεται. Αυτό είναι ένα πρόβλημα λοιπόν και γι' αυτό θα ήθελα να παραμείνουμε στο αρχικό κείμενο. Τώρα για τα παιδιά και άλλα σημαντικά θέματα θα πρέπει να υπάρχει όντως επαφή, επαφή με τους γονείς ή τους και δαιμόνες. Επίσης υπάρχει μια άλλη ε, διάταξη που μιλά για ανθρώπους με αναπηρίες. Στην πράξη όμως συχνά οι άνθρωποι αυτοί παρενοχλούνται και παραβιάζονται και τα δικαιώματά τους συχνότερα. Γιατί είναι εύκολη στόχη για του υπερβολικούς ε, ε, αστυνομικούς. Ε, γι' αυτό θα ήθελα να ληφθεί υπόψη και αυτό το πρόβλημα και ε, να επαναλαβώ τις ευχαριστήσεις μου για μια, ένα εξαιρετικό νομοθέτημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Gratuláljak a jelentéstevőnek kiváló munkájához és kompromisszumkészségéhez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 θα ε, πρόκειται για μια απτή εγγύηση για τους ε, πολίτες, πρόκειται για μια οδηγία πολύ σημαντική για την Ευρώπη χωρίς σύνορα. Τι συμβαίνει, μπορώ να ξαναρχίσω. Υπήρξε κάποιο πρόβλημα στο σύστημα διερμηνίας. Η κυρία Γκάλ. Σας ευχαριστώ. Έλεγα ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική οδηγία για την Ευρώπη, ε, μια Ευρώπη χωρίς σύνορα, όπου η ελευθερία κυκλοφορία των ανθρώπων, των κεφαλαίων και των εμπορευμάτων ε, Εξαρτάται και από την καλή γνώση των διαδικασιών από πλευρά των πολιτών και οι πολίτες θα πρέπει να χαίρουν τη στήριξη ε, ενός δικηγόρου κατά τη διάρκεια ποινική διαδικασίας αλλά να μπορούν να έχουν και επαφή με τους ε, δικούς τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξουν διαδικαστικές εγγυήσεις διότι αυτές ακριβώς οι εγγυήσεις θα δώσουν σάρκα και οστά στους στόχους της ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρομέρο, η κυρία Ρομέρο, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ως σκιώδης εισηγήτρια των σοσιαλιστών για την οδηγία αυτή θα ήθελα σήμερα να ε, τονίσω το εξής. Αύριο θα ψηφίσουμε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του, της δέσμης των δικονομικών εγγυήσεων ε, οι οποίες είχαν ξεκινήσει κατά τη διάρκεια της Σουηδικής Προεδρίας. Είναι επίγοντα όλα αυτά για να γίνουμε ένας χώρος πραγματικά ε, δικαιοσύνης. Ε, το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης είχε ως στόχο τη δημιουργία μιας ασφαλούς Ευρώπης. Με αυτή την οδηγία καθιστούμε εφικτή ε, και την δίκαιη Ευρώπη πέρα από την ασφαλή. Παλέψαμε σε αυτή την οδηγία οποιοδήποτε να έχει πρόσβαση σε δικηγόρο από τη στιγμή που θα υπάρχουν υποψίες για το πρόσωπό του χωρίς ακόμα να έχει κατηγορηθεί επισήμως. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Αντωνέσκου, τις υπόλοιπες προεδρίες, ε, τους σκιώδεις εισηγητές, διότι ε, καταφέραμε να φτάσουμε σε ένα πολύ συνενετικό αποτέλεσμα. Ε, είναι μια οδηγία η οποία ενισχύει τις εγγυήσεις στον πολίτη, δεν είναι μια οδηγία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Το δικαίωμα πρόσβασης βέβαια δεν θα είναι πραγματικότητα για όλους, διότι η Επιτροπή δεν θέλησε, δεν να ε, προβλέψει μια διάταξη ε, κατοχήρωσης του δικαιώματος πρόσβασης σε δικηγόρο όταν ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος δεν έχει τα δικά του οικονομικά ε, μέσα άρα μόνο οι ύποπτοι που μπορούν να το πληρώσουν αυτό το δικαίωμα μπορούν να το απολαύσουν. Οι ευάλωτε και οι ανήλικοι ε, δεν περιλαμβάνονται εδώ και ελπίζουμε αυτές οι ελλείψεις να διορθωθούν λίγα συντόμως. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Ρομέρο. Και τώρα δίνω το λόγο στην κυρία Μακοβέη για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Είναι όντως σημαντική η πρόσβαση σε δικηγόρο αμέσως μετά τη σύλληψη ε, κάποιου. Αυτό είναι ζωτικό ε, στοιχείο της ισονομίας, της ε, ίσης διαδικασίας. Μιλούμε για το άρθρο 6 της Σύμβασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο προβλέπει ότι η δίκη πρέπει να είναι δίκαιη και να έχει κατοχυρωθεί το δικαίωμα στην υπεράσπιση σε πολλές ε, περιπτώσεις λοιπόν αυτό το δικαιώμα έχει καταστρατηγηθεί. Πέραν όλων αυτών όμως η υπεράσπιση θα πρέπει να είναι αποτελεσματική, να είναι ουσιαστική, να υπάρχει αληθινή υπεράσπιση. Ο οποίο δεν μπορεί να πληρώσει δικηγόρο σε μια ποινική διαδικασία, ε τότε θα πρέπει το κράτος να του προσφέρει έναν δικηγόρο. Και υπ' αυτή την έννοια καταφέραμε να μπει αυτό το δικαίωμα στη δικαστική ε, δωρεάν συνδρομή αρρωγή για όσους δεν έχουν αυτά τα μέσα στη διάθεσή τους. Και είναι και πολύ σημαντική η υπεράσπιση προμπόνο. Θα πρέπει οι δικηγόροι να συμβάλλουν και να προσφέρουν ε, αυτό το σημαντικό βοήθημα στην κοινωνία. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ε, Κινούμε τώρα τη διαδικασία ΚΑΤΣΤΙΑΙ. Ο κύριος Διαθεμέρα. Κύριε Πρόεδρε, η ποινική διαδικασία ενισχύεται με αυτή την οδηγία. Έχουμε περισσότερες εγγυήσεις, περισσότερη δικαιοσύνη, περισσότερη ποιότητα. Οι ύποπτοι και οι κατηγορούμενοι θα έχουν δικηγόρο από τα αρχικά στάδια της ε, διαδικασίας, ανεξαρτήτως ε, εάν τους έχει επιβληθεί κύρωση στερητική της ελευθερίας ή όχι. Και θα ο δικηγόρος θα μπορεί να λαμβάνει γνώση όλου του φακέλου και δεν θα υπάρχουν ε, περιορισμοί στην <laughs> συχνότητα και στη διάρκεια ε, των συναντήσεων του κατηγορημένου ή του υπόπτου με τον δικηγόρο του και μάλιστα κατηδίαν. Το πιο σημαντικό είναι αυτό το ακριβώς το γεγονό ότι η επικοινωνία υπόπτου, κατηγορουμένου και δικηγόρου γίνεται απολύτως κατηδίαν ε, θα υπάρχει πλήρη εμπιστευτικότητα και πλήρε απόρριτο. Θέλω να συγχαρώ την κυρία Συγήτρια, την κυρία Αντωνέσκου για την καταπληκτική της δουλειά η οποία ε, δόθηκε και ψυχή και σώμα σε αυτόν τον αγώνα προκειμένου να καταλήξουμε σε αυτή την τόσο, σε αυτό το τόσο σημαντικό ε, κείμενο. Θέλω να ευχαριστήσω όλους λοιπόν όσοι έχουν συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ ο κύριος Ιντάλγο. Ως δικηγόρος, έχοντας ασκήσει το επάγγελμα τέσσερις δεκαετίες, χαιρετίζω το τόσο σημαντικό βήμα που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Η οδηγία αυτή όμως δεν περιλαμβάνει το δικαίωμα ε, πρόσβαση στη δωρεάν δικαιοσύνη, κάτι το οποίο προβλέπεται μόνο στην εθνική νομοθεσία, δυστυχώς και αυτό πρέπει να το παραδεχθούμε. Στην Ισπανία, παρόλο που ο υπουργό αυτή τη στιγμή δεν είναι ένθερμος οπαδός αυτού του θεσμού που έχουμε προβλέψει, έχουμε την ε, δωρεάν υπεράσπιση και δικαστική ε, συνδρομή ε, και Εάν όλα αυτά τα επιταχύνουμε, τα αποτελέσματα θα είναι ακόμα καλύτερα. Θα μπορούσαμε, ας πούμε, να κατευθύνουμε τους νέους δικηγόρους ε, προς αυτή την κατεύθυνση ε, και αυτό θα οδηγούσε σε ένα χώρο περισσότερης ελευθερίας και δικαιοσύνης για όλους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπιλμπάου για ένα λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και θέλω να ευχαριστήσω και την κυρία Αντωνέσκου για όλη αυτή τη δουλειά που έχει κάνει. Οι οδηγίε που έχουν να κάνουν με τα ποινικά συστήματα των κρατών μελών είναι περίπλοκε, αλλά συμβάλλουν στη βελτίωση τη προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η οδηγία θα θυμίσει στου πάντε ότι το Ευρωπαϊκό το Δικαστήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα δεν θεωρεί ότι ισχύουν τα αποδεκτικά στοιχεία που έχουν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια ανάκρισης χωρίς παρουσία δικηγόρου και θα πρέπει να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην ε, ε, νομική υπεράσπιση. Θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα ε, βήματα για να καταπολεμήσουμε και το οργανωμένο έγκλημα. Όλες αυτές οι εξαιρέσεις έχουν οδηγήσει σε περισσότερες περιπτώσεις βασανιστήριων. Αυτό ισχύει και με, στη βασκική αστυνομία της Έντσα. Θα πρέπει να συντονιστούν καλύτερα οι αστυνομίες της Ευρώπης. Κύριε Ρέντιν, θα πρέπει αυτό να το καταγράψετε ως καλή πρακτική την οποία θα πρέπει να μοιραστείτε με τις υπόλοιπες αστυνομικές δυνάμεις της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπρόν σε ένα λεπτό. Ίσως αυτό να μην ε, ισχύει ακόμα στην ε, Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά υπάρχουν σημεία ανησυχία. Το ουσιαστικό περιεχόμενο είναι όντω ε, σωστό. Θα πρέπει οποιοδήποτε ύποπτο να χαίρει όλων αυτών των δικαιωμάτων. Ωστόσο δεν χρειάζεται ευρωπαϊκή νομοθεσία. Μια τέτοια νομοθεσία δεν αντιστοιχεί, δεν ικανοποιεί απόλυτα τι ανάγκε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ακόμα ολόκληρο ο κόσμο κόσμος ε, και ο κόσμος που ε, ταξιδεύει δεν περιορίζεται μόνο στα κράτη-μέλη. Δεν χρειάζεται ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά μια διεθνή συνθήκη που θα περιλαμβάνονται και θα συνυπογράφουν όσο γίνεται περισσότερες χώρες στον κόσμο, ώστε αυτά τα δικαιώματα να εφαρμόζονται σε όλες αυτές τις χώρες. Εγώ έχω το αίσθημα πως αυτή η πρόταση δεν αφορά τόσο τα δικαιώματα των υπόπτων ε, μέσω της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, αλλά αφορά περισσότερο την επέκταση των ευρωπαϊκών ε, νομοθετικών ε, αρμοδιοτήτων και το θέμα είναι μόνο ένα μέσο για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος της Επιτροπής θα δώσω το λόγο στην κυρία Ρέντινγκ. Πρόεδρε, υπάρχει σχεδόν ομοφωνία στο σώμα πως πραγματικά κάνουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Δικαιοσύνης σε, ολόκληρο, σε όλα μας τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας σε ολόκληρο το Κοινοβούλιο, σε αυτή τη διαδικασία συναπόφασης ε, που μας βοήθησε να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Επιτύχαμε πολλά, αλλά πρέπει να γίνουν κι άλλα. Πολύ Ήδη αναφερθήκατε στο επόμενο βήμα που όπως σας είπα θα έρθει, θα γίνει μέσα στο φθινόπωρο. Ε, θα είναι μια δέσμη πρωτοβουλειών για ειδική, ε, ειδική προστασία των παιδιών, νομική αρρωγή και το τεκμήριο αθότητας. Ε, αν όλα αυτά προσθεθούν σε ολόκληρη τη δέσμη που ήδη έχουμε αποφασίσει, μπορούμε πραγματικά να πούμε ότι ότι πραγματικά δουλέψαμε υπέρ της δικαιοσύνης για την Ευρωπαϊκή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα δίνω το λόγο στην συγχύτρια την κυρία Αντωνέσκου. Ευχαριστώ πολύ. πολύ καλή η συζήτηση που κάναμε σήμερα το απόγευμα και σας ευχαριστώ πολύ. Στη δουλειά που κάναμε για το θέμα αυτό με τους χιώδης εισηγητές, πάντοτε ο στόχος μας ε, ήταν ε, να λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα ε, των κατηγορημένων και υπόπτων, αλλά παράλληλα είχαμε υπόψη μας και το κοινό καλό, ούτως ώστε να έχουμε μια καλή διαχείριση στο επίπεδο των διοκτικών αρχών. Κάθε οδράσεις ε, ε, θα πρέπει ε, να την χάνει των απαιτούμενων κυρώσεων αναλογικά προς, το, προς την αξιόπινη πράξη που έχει διαπράξει και αυτό προσπαθήσαμε να εξασφαλίσουμε μια εξισορρόπηση του χώρου ασφάλειας Ελευθερίας και Δικαιοσύνης. Ε, χαιρετίζω αυτά τα οποία μας ανέφερε η κυρία Ρέντινγκ για το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για τους επόμενους ε, μήνες ε, και για τα δικονομικά δικαιώματα. Θέλουμε εγγυήσει ε, για τους υπόπτους ε, και ε, τους κατηγορουμένους σε επίπεδο δικαστικής αρρωγής και παροχής νομικών συμβουλών. Πιστεύω ότι αυτά είναι σημαντικά μέτρα στο, στη δέσμη αυτών των μέτρων. Ελπίζω λοιπόν ότι το συντομότερο δυνατόν θα μπορέσουν να υλοποιηθούν αυτά τα μέτρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Αντωνέσκου. Και θα ήθελα και εγώ να σας συγχαρώ όπως και οι άλλοι συνάδελφοι και κλείνω με δύο παρατηρήσεις. Η κυρία Λάτφορντ είπε ότι